παίξει. Σας ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας με την έκθεσή σας και αναμένουμε να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε πώς θα έχουμε τις κατάλληλες πολιτικές. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί αύριο. Τελευταίο σημείο για σήμερα είναι η έκθεση Κοτσολίνο για την καταπολέμηση της απάτης. Για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Κοτσολίνο. Presidente, in un momento in cui il Trattato di Lisbona rende più incisivo il ruolo dell'Europa nella vita di milioni di cittadini. Στη φάση της υλοποίησης της συνθήκης της Λισαβόνας που δίνει παραπάνω δικαιώματα στους πολίτες η πρόκληση που έχουμε για την καταπολέμηση της απάτης είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εμείς έχουμε το σενάριο που του 2008 του ελεγκτικού συνεδρίου όπου δια όπου διαπιστώνουμε μία μείωση της απάτης από το 2007 στο 2008. Όμως οι απόλυτες τιμές δεν μας δείχνουν πού βρίσκεται η κατάσταση, πού είναι άσχημη και πού ελέγχεται. Εμείς λοιπόν δίνουμε προτεραιότητα σε δύο πράγματα. Πρέπει να υπευθυνοποιηθούν παραπάνω τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των παρατυπιών. Να διαδίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες να καταγγέλουν απάτες. Επίσης πρέπει να ξεκινήσουμε με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη δυνατότητα παρέμβαση των κρατών μελών με στρατηγικές και διοικητικές διαδικασίες που θα έχουν ως επίγγελμα την πρόκειται του σχεδίου και που θα έχουν επιπτώσει στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Για να προσθέσουμε αυτούς τους στόχους στο Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει σε προτεραιότητες όπου η Όλαφ θα πρέπει να φτιάξει 27 δελτία για το κάθε κράτος μέλος και όπου θα αναφέρονται με συγκεκριμένη χαρτογράφηση οι απάτες και οι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν στην κάθε χώρα, αυτοί που γίνονται και η ποιότητά τους. Δεύτερο, να μειωθεί η απάτη βελτιώνοντας τους κανονισμούς. Απλούστευση νομοθετική απλούστευση και ρυθμιστική απλούστευση για τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης, θα πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα κατά της ε, χρηματοπιστωτικής απάτης και της τρέβλωσης των δημοπρασιών. Αυτά είναι... Αυτά τα συμμερίζεται και η Κομισιόν. θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με τους φορολογικούς παραδείσους που διαφεύγουν τα κεφάλαια. Χρειάζομαστε λοιπόν στρατηγικές κατά της απάτης και κατά της διαφθοράς. Στο τέλος για την Όλαφ θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητη στη λειτουργία της από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να έχει και το επαρκές προσωπικό. και θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για μια ενιαία ευρωπαϊκή εισαγγελία. Πρέπει να παλέψουμε από κοινού για τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε χειραγώγηση, να δώσουμε τα απαραίτητα μέσα στην υλοποίηση του κοινοτικού σχεδίου. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι στρεβλώσεις ε, στις, ε, στα κοινοτικά οικονομικά και να κάνουμε βήματα προς τα μπρος βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης. Πιστεύω ότι αν καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα θα πετύχουμε να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καλύπτει και τις απαιτήσει των πολιτών. Κάτσε. the Η κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ως κοιόδης του ΕΛΚ θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή και στους άλλους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Θέλουμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια και καλύτερους κανόνες δημοσίων προμηθειών γιατί εκεί βρίσκεται το επίκεντρο των απατών και της διαφθοράς. Επίσης, οι δικαιούχοι κοινοτικών κονδυλίων θα πρέπει να φαίνονται σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Επίσης, η πέτη απάτης δεν θα πρέπει να είναι στελέχη επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει οι εθνικές αρχές να προβάλλουν αγωγές με βάση τα δεδομένα της ΟΛΑΦ γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δρούν σε υπεράκτια συστήματα. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει την απάτη και τη διαφθορά σαν θέμα ε, άμεσης προτεραιότητας. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλη. Δεν ε, είναι υπερβολικό να πούμε ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι απότοκη μίας ηθικής ε, κρίσης. Δυστυχώς ε, επικρατεί η απάτη και η διαφορά κατά της αλληλεγγύης και μέχρι ότι φτάσουμε στην γενοδορία και την αλληλεγγύη δεν θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη με κάθε μέσο. Στην Ιρλανδία αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα και στη Βόρειο Ιρλανδία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βεβαίως οι τράπεζες είναι η βασική υπέτη γιατί δεν λογοδοτούν. Αυτό μας οδήγησε σε μεγάλα προβλήματα στην Ιρλανδία και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι απάτες να σταματήσουν και οι υπέτοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Ο Επίτροπος, κύριε Ντάλη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, εξ του συναδέλφου του Επιτρόπου Σεμέτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική του έκθεση, για την ε, προώθηση των χρηματοοικονομικών μας συμφερόντων. Η Κομισιόν εκτιμά το ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει κοινή ευθύνη όλων των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σε σχέση ε, με την ε, ε, απόδοση ευθυνών. Η Όλαφ έχει προβεί στη σύσταση ενός νέου συστήματος IMS μία νέα μορφή διαχείρισης έτσι ώστε να καταγράφονται οι παρατυπίες των κρατών μελών όπως επικρίνονται στην έκθεση σας. Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν μεγάλη σημασία και μας απασχολούν και στην Κομισιόν. Εμείς προσπαθήσαμε να καταπραίνουμε αυτές τις αδυναμίες στις πληγήσεις περιοχές και τομείς μέσα στα πλαίσια του 2008 με μια διαδικασία απλοποίησης. Μαζί με τον Επίτροπο ΣΕΜΕΤΑ θα προωθήσουμε αυτή τη δράση έτσι ώστε να προωθήσουμε μια πολιτική σύνοχης και θα, θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για το κλείσιμο των προγραμμάτων του 2008 και στη νέα περίοδο προγραμματισμού θα ευεργετηθούν τα κράτη-μέλη. Επίσης, θα συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές έτσι ώστε να ε, υπάρξει πλήρης ανάληψη ευθυνών όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδος ως προς τη διαφάνεια των ε, ευεργετηθέντων και θεωρούμε ότι οι δικαιούχοι, το θέμα των δικαιούχων αφορά τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει μία ιστοσελίδα ανά κράτος μέλος με βάση την επιμερισμένη ευθύνη. Για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση θα υπάρχουν ειδικά ε, links για αυτές τις ιστοσελίδες. Τώρα ως προς την ε, Όλαφ. Θεωρώ πως πρέπει να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη στήριξη του έργου του Όλαφ ο συναλφός μου, ο κύριος Σεμέτα, συμφωνεί απολύτως πως η υπηρεσία πρέπει να επικεντρωθεί στα βασικά καθήκοντα, δηλαδή τις έρευνες, παρά το ότι έχει και άλλα σημαντικά καθήκοντα. Ο Όλαφ, ειδικά στον τομέα της πρόληψης απάντησε. Επίσης συμφωνεί πως πρέπει ο Όλαφ να δώσει βάρος πιο σημαντικές περιπτώσεις και οι μικροαπάτες να απασχολήσουν άλλους φορείς. Το 2008 αναθεώρησε τις διαδικασίες ε, δημοσιονομικής παρακολούθησης με το να ορίσει κάποια όρια επιέλατων. Ο κύριος ε, Σεμέτα σημειώνει το ότι πρέπει να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Ο Όλαφ επίσης, ο Όλαφ και ο IAS συνεργάστηκαν στενότατα από το 2003, ανταλλάσσουν πληροφορίες και υπάρχει εκπαίδευση για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντο. Ο Όλαφ είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί ακόμη στενότερα με το IAS όσον αφορά τα, δικαι... τα δικονομικά δικαιώματα. Ο νέος κανονισμός του Όλαφ του 2009 προβλέπει το τι πρέπει να κάνουν οι ερευνητέ του Όλαφ. Πιο λεπτομερεί κανόνες για αυτά τα δικαιώματα θα συμπεριληφθούν στην νομοθετική πρόταση περί αναθεώρησης του κανονισμού του Όλαφ. Η Κομισιόν θέλει εδώ πέρα να υπενθυμίσει πως υπάρχει ένα έγγραφο προβληματισμού για τη μεταρρύθμιση του Όλαφ που θα πάει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζουμε λοιπόν να τα παρουσιάσει ο Επίτροπο στην, ε, επιτροπή του, στην συνάντηση με την Επιτροπή Προπολογισμού τον Ιούλιο και θεωρεί πω το Κοινοβούλιο είναι σύμμαχο στον αγώνα μαζί με τον Όλαφ για την προστασία των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το θέμα αυτό θα ψηφιστεί αύριο. Η κυρία Μπασέσκο και πάλι. Θα ήθελα να συμπεριλευθεί η ομιλία μου για την καταπολέμηση της απάτης στην Ολομέλεια γιατί Ίσως ε, θεωρείτε ότι το ένα θέμα σχετίζεται άμεσα με το άλλο. Ναι, θα συμπεριληφθεί η ομιλία σας. Θα συμπεριληφθεί σε αυτό το σημείο της ημερής διάταξης και όχι στο προηγούμενο.